Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως, λέει ο κύριος Σάσολη. Και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, έχουμε πρώτα την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιδημία.